εξονόματος προς τους Σύρους πρόσφυγες. Ο κύριος Δελαβέτοβα, πρώτος εξονόματος του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οφείλει να είναι λέγει και η ε, δική μας η Προεδρία τα ενισχύει όλα αυτά. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο τους ε, προσέφεραν 1,5 δις ευρώ στη μορφή οικονομικής βοήθειας όταν ξέσπασε η κρίση στη Συρία το 2011. Και σε αυτά προστίθενται τα 600 περίπου εκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας που προήλθαν από τον προεπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εκταμιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ξέρουν πολύ καλά οι ευρωβουλευτές, μόλις ε, ε, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός ο διορθωτικός του 2014 που προβλέπει άλλα 200 τόσα περίπου εκατομμύρια για την ανθρωπιστική βοήθεια εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφέτος. Ένα μεγάλο τμήμα αυτού του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συριακή κρίση. Αυτό λοιπόν είναι μια σαφής ένδειξη του πόσο είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που του χρειάζονται, κυρίως σε αυτούς που έχουν πληγεί από την κρίση στη Συρία. Εχθές το Συμβούλιο ανέκρινε τα συμπεράσματά του για την κατάσταση στη Συρία. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας ανησυχία για το ότι δεν υπάρχουν κονδύλια ε, μετά από την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για το 2014 και έτσι λοιπόν σταμάτησε η προσωρινή βοήθεια προς τους Σύριους πρόσφυγες από πλευράς επισητιστικού παγκόσμιου επισητιστικού προγράμματος. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τη χρηματοδότηση ε, λόγω του χειμώνα και ε, μετά από τις εκκλήσεις που έχουν γίνει για το 2015. Όμως δεν ζητήσαμε μόνο από τους άλλους βοήθεια. Ε, τα κράτη-μέλη είναι βασικοί δωρητές που αντέδρασαν πάρα αυτά. Όσον αφορά ε, την ε, επίκληση του World Food Program για την ε, χρηματοδότηση για τη Συρία, ας πούμε η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο από κοινού συνεισέφεραν πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια. Έχουμε λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίδει μια συλλογική απάντηση σε αυτή την έκκληση για πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Χαιρόμεθα πάρα πολύ που με τον τρόπο αυτό κατορθώσαμε πλέον να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις που υπήρχαν στο Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα και ε, το 1,7 εκατομμύρια πρόσφυγες μπορούν πλέον να ε, βοηθηθούν. Παραμένει τραγικό το γεγονός ότι μια κρίση όπως αυτή στη Συρία, μια τέτοια κρίση δυστυχώς ε, δεν ε, βρίσκει ανταπόκριση για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των εκτοπιστέντων. Πολλοί εξ αυτών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Συρία και αυτό το έκαναν φεύγοντας και παίρνοντας μαζί τους μόνο τα ρούχα που φορούσαν. Μπορούμε βέβαια ε, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αυξηθεί περαιτέρω ο πόνος τους, να τους βοηθήσουμε επισητιστικά σε αυτούς που έχουν χάσει τα πάντα γιατί κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου λοιπόν συντονίσαμε πάρα πολύ προσεκτικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μέσα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απάντησή μας σε αυτή την κρίση χωρίς προηγούμενο. Ε, θέλουμε να υπάρχει μια συλλογική απάντηση και να προσπαθήσουμε στο βαθμό του δυνατού να ε, καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην παγκόσμια χρηματοδότηση. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τους βασικούς δωρητές του World Food Program και μετά από την πρόσφατη έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν 150 περίπου εκατομμύρια ευρώ ε, για, με τη μορφή βοήθειας για την κρίση στη Συρία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το ε, πρόγραμμα της επιστηστικής βοήθειας είναι απαραίτητο για να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ως κρατη σε διμερή βάση έχουμε μία μακρά παράδοση συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν... Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τόσο για τη χρηματοδότηση όσο και για τον προγραμματισμό. Οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι ελλείψεις που προέκυψαν κατά παρελθόν δεν θα προκύψουν στο μέλλον. Οφείλουμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα, κυρίως τους αθώους άμαχους αυτού του τραγικού, του ολέθριου πολέμου στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ Δελαπέτο, και σας ευχαριστώ Επίση, που λάβατε υπόψη ότι έχουμε πρόβλημα χρόνου. Τώρα εξ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο του κ. Στυλιανίδη, παρακαλώ. Very much, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό το σημαντικό θέμα σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση στη Συρία είναι χωρίς προηγούμενο και σε επίπεδο ανθρωπιστικών συνεπειών αλλά και σε επίπεδο οικονομικών συνεπειών. Μια άμεση αντίδραση των διεθνών δωρητών είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να ε, μην χειροτερεύσει περαιτέρω η κατάσταση. Μια ε, πλήρης απάντηση στην κρίση δεν μπορεί να καλυφθεί από τους κανονικούς μας προϋπολογισμούς. Πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να υπάρξει όμως μια ισχυρή ανταπόκριση. Έχουμε συλλογική ευθύνη να βρούμε τους στόχους για να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Οι αποφάσεις για μειώσεις της βοήθειας σε τρόφιμα δείχνουν το πόσο οικονομικά επιβαρημένη είναι η κατάσταση μετά από αυτήν την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ανταποκρίνεται βέβαια στις ανάγκες της κρίσης στη Συρία. Ανταποκρινόμεθα στην έκκληση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να ε, υπάρξει εκ νέου ε, βοήθεια προς τους ε, Σύρους πρόσφυγες. Θα ήθελα εγώ να εκφράσω την ε, ε, ικανοποίησή μου για την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η γέτιδα. Έχουμε δώσει πάνω από 2 δις ευρώ από αυτά τα 600 εκατομμύρια, 621 εκατομμύρια προέρχονται από τον προϋπολογισμό ε, για τα ανθρωπιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 132 εκατομμύρια δόθηκαν στις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Συρία και στις γειτονικές χώρες. Ο παγκόσμιο αυτό επισητιστικό πρόγραμμα είναι ε, το δεύτερο μετά από την Οργάνωση για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς συνεχίζουμε την εμπλοκή μας με τον Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα. Κατεπηγόντως δώσαμε επιπλέον 5,5 εκατομμύρια ευρώ για τους Σύρους πρόσφυγες. Με το ποσό αυτό η χρηματοδότηση την οποία δίδουμε για το 2014 θα φτάσει τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Συν φυσικά τα 61 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2013. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, θα κινητοποιήσουμε και επιπλέον πόρους. Δεν είναι τυχαίο το ότι εδώ και λίγες μέρες και το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα και η Βάλερη Άμος ε, εξέφρασαν ε, την ε, εκτίμησή τους για την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι αλήθεια ότι το παγκόσμιο επισητιστικό πρόγραμμα έχει μακράν τις μεγαλύτερες ανάγκες που θα φτάσουν περίπου στο 1,8 δις δολάρια φέτος. Το ποσό αυτό ξεπερνά το 1,6 δις δολάρια που ε, δίδε, βοήθεια που δίδεται στην οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Μόνο το 60% των αναγκών αυτών καλύπτεται από, τις, από τα διαθέσιμα. Δυστυχώς ε, το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα είναι ένας μόνο από τους εταίρους μας που έχουν τεράστιες τραγικές ανάγκες οικονομικά. Γι' αυτό έχουμε πει εμείς προς την κοινότητα των δωρητριών χωρών ότι τα κενά που υπάρχουν στην χρηματοδότηση δεν είναι βιώσιμα. Η Συρία είναι η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά δεν είναι η μόνη κρίση. Έχουμε το Ιράκ, την κεντροαφροκανική Δημοκρατία κτλ. Όλες αυτές οι κρίσεις έχουν ναι, πράγματι εξαντλήσει τους ε, ανθρωπιστικούς προϋπολογισμούς. Τα χρήματα ποτέ δεν θα φτάνουν βέβαια, ως εκ τούτου απαιτείται μια πιο αποτελεσματική ε, παρέμβαση σε επίπεδο κόστους. Αυτό ισχύει επίσης και για το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα. Φέτος 165 εκατομμύρια θα έχουμε δώσει ε, για τον προϋπολογισμό. Λιγότερα από τα έκτακτα 300 εκατομμύρια τα οποία κινητοποιήσαμε το 2012. Τον επόμενο χρόνο ο αρχικός ε, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια και θα ε, υπάρξουν όμως νέοι πόροι σύντομα. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και τους μοχλούς που έχουμε για να το πετύχουμε. Οι προσπάθειές μου όμως ε, από μόνος μου δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν αρκούν. Απαιτείται ισχυρή συλλογική δράση για τον επόμενο χρόνο. Ε, αναμένουμε ανάγκες 7,2 δις δολάρια για την κρίση στη Συρία μόνον. Πρόκειται για μια τεράστια αύξηση σε σχέση με τα 6 δις που χρειάστηκαν το 2014. Η Συριακή κρίση είναι η βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Το σύνολο της περιοχής ε, υποφέρει από την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους αύξησης της χρηματοδότησης και επίσης θα πρέπει να καταστήσουμε τη χρηματοδότηση αυτή βιώσιμη. Αλλιώς θα είναι ένα μπάλωμα στην κατάσταση. Πρέπει να συνεχίσουμε εμείς ε, να τιμάμε τις υποχρεώσεις μας. Το θέμα δεν είναι μόνο το ηθικό μας καθήκον, αλλά είναι θέμα ζωής και θανάτου για εκατομμύρια προσφύγων στη Συρία. Όπως ξέρετε πριν λίγες μέρες επανήλθα από μια κοινή αποστολή με την κυρία Μογκερίνη και τον Επίτροπο Χάν στην Τουρκία. Εκεί επισκεφθήκαμε ε, και ε, καταλήματα προσφύγων στο νότο της Τουρκίας. Η κατάσταση είναι πραγματικά ιδιαίτερα κακή και αν μειωθεί η βοήθεια για την αγορά τροφίμων είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα. Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση. Τελικά, αυτό το οποίο χρειάζεται για την κρίση της Συρίας βέβαια είναι μια πολιτική λύση. Ο κύριος Στούρα ο εκπρόσωπος των ειδικό απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζεται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό φάνηκε χθε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Σιλιανίδη, αγαπητοί συνάδελφοι ακολουθεί συζήτηση. Δυστυχώ έχουμε ακόμα περισσότερη καθυστέρηση και θα είμαι αρκετά αυστηρό και παρακαλώ την κατανόησή σα. Πρώτο ο κύριο Στυρ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την τελευταία τετραετία από τότε που άρχισε η ένοπλη σύνταξη στην Συρία επανειλημμένα τονίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση σήμερα παγκοσμίω. 14 ε, εκατομμύρια ε, χρειάζονται οπωσδήποτε βοήθεια και είναι παιδιά τα περισσότερα. 1,7 εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες που ε, εποφελούνται από το ταμείο, αυτό το παγκόσμιο επισκεπτιστικό ταμείο. Αλλά τώρα κόπηκαν τα κονδύλια. Θα πρέπει το συντομότερο να επανέλθουν στο Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα. Είναι ενθαρρυντική η αντίδραση του κυρίου Στυλιανίδη γιατί ανακοινώνει οικονομική βοήθεια. Θα πρέπει να τονίσουμε οπωσδήποτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να τηρήσει όλες τις υποσχέσεις ε, εγκαίρως γιατί ακούμε και παράπονα ε, εμείς εγκαίρως λοιπόν καταβάλουμε τα κονδυλία, αλλά θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή για χώρες όπως τη Συρία. Εδώ ε, εξαρτώνται από τη βοήθεια αυτή οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι διεθνείς εταίροι που θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ανθρωπιστική κρίση στη Συρία χρειάζεται πολιτική λύση αν δούμε τι ρίζες και τι αιτίε. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε τι προσπάθειές μα. Ευχαριστώ πολύ. Να πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Στυρ Και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Νόιζε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αξιότιμη Υπουργέ, όλοι οι πολιτικοί θέλουν γρήγορα να βρεθεί πάρα πολύ βοήθεια για τους σύρους πρόσφυγες, αλλά το Ταμείο είναι μείον το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και γίνονται οικονομίες και για τα τρόφιμα. Είναι ε, σαφής η στάση των πολιτικών που με πάθος προειδοποιούν ε, από το θάνατο και τα δεινά. Ένα παράδειγμα. Ε, η γερμανική κυβέρνηση, στην οποία ανήκει και το κόμμα μου, είπε ότι είναι η καταστροφή του αιώνα. Σωστά το ακούστε, του αιώνα. Βρέχει. Ε, ε, μετά ε, έρχεται το ψύχος και ο θάνατος τελικά. Ε, περισσεύει η δραματουργία και η συμπόνια. Αλλά τι νόημα έχει όλο αυτό το πάθος και η δραματουργία εάν η νυφαλιότητα των αριθμών δεν ανταποκρίνεται. Γιατί οι αριθμοί είναι γυμνοί και σαφείς. Ο προπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια από το 2013 συνεχώς ερικνώνεται χρόνια η κατάσταση και σκεμένα υποχρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη. Ε, και έχουμε και πάλι απλήρωτους λογαριασμούς, τους οποίους ε, φέρνουμε και τους μεταφέρουμε από το ένα έτος στο άλλο. Και το λέω όχι επειδή έρχονται Χριστούγεννα, να ανοίξουμε και τις πόρτες μας και τα σύνορα και τις καρδιές μας, αλλά τα κράτη-μέλη να ανοίξουν την τσέπη τους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Κάσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μία από τις πιο αιμοσταγείς σειράξεις τελευταίας δεκαετίας είναι αυτή που σοβεί ε, στην Συρία. 200.000 ε, έχουν φτάσει οι νεκροί και πάρα πολλοί είναι εκτοπισμένοι. Βλέπουμε περιοχές που μιλούσαν αραμαϊκά, που είναι η γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός και ε, ε, οι άνθρωποι αυτοί δολοφονούνται, διώχνονται από τις αιστείες τους, ε, αφανίζονται. Χιλιάδες πρόσφυγες φεύγουν προς άλλες χώρες, εκτός από τους εκτοπισμένους εντός της Συρίας και είναι πολλοί και οι ανήλικοι. Είναι τραγωδίες αυτές προσωπικές, οικογενειακές, τεράστιες και τον τελευταίο μήνα Δυστυχώς έχει σταματήσει η χρηματοδότηση από το επιστημιστικό πρόγραμμα. Ε, το πρόγραμμα αυτό που έπρεπε να είναι εγγύηση ε, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει ε, τα ποσά που είχαν υποσχεθεί. Και επίσης σας παρακαλώ, σας κλιπαρώ. Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Τέλιτσκα. Uh, uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Έχουμε μια συνάντηση της ομάδας για ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητάμε αύριο θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή. Ανταποκρίθηκε γρήγορα και με επάρκεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά παραμένει η ανησυχία. Νομίζω ότι η διακοπή της βοήθειας σε ε, τρόφιμα δεν είναι μόνο κάτι το βλαβερό. Είναι σχεδόν ένα έγκλημα ε, βλέποντας ε, ε, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρόσφυγες. Σε λίγους μήνες ε, θα εξακολουθούμε να έχουμε δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα. Το συνειδητοποιείτε κύριε Επίτροπε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω να είστε σκληρός. Ακούγεται σαν κλισέ αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι θα σας στηρίξουμε να είστε έντονος, να είστε απαιτητικός προς τους εταίρους μας. Το θέμα δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες, είναι και η κατάσταση στις γειτονικές χώρες όπου καταραίουν τα συστήματα της οικονομίας, τα κοινωνικά συστήματα, τα τρόφιμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Λίβανο. Ε, στα 4 εκατομμύρια πάνω από 1 εκατομμύριο είναι πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι τραγική πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί για το θέμα αυτό. Θα σας στηρίζουμε στο μέλλον, αλλά έχουμε και προσδοκίες υψηλές από σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Χρυσόγονος, παρακαλώ. Στη Συρία έχει αναγκάσει πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλες χώρες, πολλοί από αυτούς σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έκκληση που απίφθινε το παγκόσμιο επιστημιστικό πρόγραμμα την 1η δεκέμβρη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους συγκεντρώθηκαν συνολικά 88 εκατομμύρια δολάρια. τα έξι από αυτά τα έβαλε η ευρωπαϊκή ένωση η οποία όμως κατά τα άλλα επιμένει στη διατήρηση των κανονισμών του δουβλίνου που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια την υγεία και την ίδια τη ζωή αυτών των ανθρώπων. το ψευδεπίγραφο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που καθιερώνουν οι κανονισμοί αυτοί είναι ένα απάνθρωπο σύστημα που παγιδεύει τους πρόσφυγες στις χώρες εισόδου δηλαδή στις μεσογειακές χώρες όπως η ελλάδα και η ιταλία οι οποίες έχουν προπολού ξεπεράσει τα όρια τους. ακόμα και η αναγνώριση της προσφυγικής τους ιδιότητας κατά προτεραιότητα δεν θα εξασφαλίσει στους πρόσφυγες αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης ούτε θα αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από τη μαζική εισρωή στις συγκεκριμένες αυτές χώρες. απαιτούμε λοιπόν ένα πιο δίκαιο σύστημα κατανομής των ευθυνών. έχει έρθει η ώρα τα κράτη της κεντρικής και βόρειας ευρώπης που είναι στην πραγματικότητα οι χώρες προορισμού των μεταναστών να δείξουν κατά πόσο ενστερνίζονται στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης που διακηρύσσουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσόγονε. Για ένα λεπτό ο κύριος Σμιθ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε. Ε, γρήγορα δράσατε μεταξύ άλλων και αντιδράσατε σε αυτή την ε, φοβερή κρίση και θα ήθελα να σας επενέσω γι' αυτό. Έχω όμως συγκεκριμένες ερωτήσεις. Υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα σε αυτό το επιστημιστικό πρόγραμμα που οδήγησε στην αναστολή της βοήθειας ή απλώς έχει κατακλειστεί από τις ανάγκες ε, και ε, υπάρχει θέμα ε, πολιτικής. Πραγματικά ήταν καταπληκτική η αντίδρασή σας, αλλά άκουσα ότι πήγατε με τους άλλους επιτρόπους στην περιοχή και είδατε και την ανθρωπιστική πτυχή που πολύ σωστά είπατε είναι ένα μόνο τμήμα. Χρειάζεται μια πολιτική λύση. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες και πληροφορίες πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίες σας ε, συντονίζονται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις ορισμένων κρατών μελών γιατί αυτό μπορεί να έχει πολλές συνέπειες και για μια συνεκτική πολιτική για τους πρόσφυγες σε ορισμένα από τα κράτη-μέλη που έχουν καλύτερες επιδόσεις πολύ συχνά κάποια κράτη από κάποια άλλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμιθ. Για ένα λεπτό ο κύριος Φουντούλης παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η αναστολή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού προγράμματο του ΟΗΕ είναι καταστροφική. Πρόσφυγε αγωνίζονται να επιβιώσουν μέσα στο χειμώνα χωρί να έχουν τα στοιχειώδη για τη σύντηση και την υγεία. Ένα εκατομμύριο 700.000 πρόσφυγες από τη συρία έχουν καταφύγει στην ιορδανία το λίβανο την τουρκία το ιράκ και την αίγυπτο. από εκεί προσπαθούν να φτάσουν στην ευρώπη που τη βλέπουν σαν τη γη της επαγγελίας. δεν μπορείς να σταματήσεις ένα πεινασμένο από την αναζήτηση τρόπων επιβίωσης. οι ηνωμένες πολιτείες εξέφρασαν την ανησυχία τους και ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα ποιο ευθύνεται όμω για την κατάσταση αυτή ποιο έφερε την πείνα και την καταστροφή στη συρία και αναγκάζει το λαό τη να παίρνει τον δρόμο τη προσφυγιά; οι μεγάλε δυνάμει που με πολεμικέ επιχειρήσει και με το πρόσχημα τη δίθεν απελευθέρωση και τη αποκατάσταση τη δημοκρατία προσπαθούν να επιβάλλουν τι πολιτικέ του. η αμερική αλλά και η ευρώπη είναι συνένοχοι για αυτή την κατάσταση όπου και να κοιτάξουμε στο ιράκ τη συρία και τη λιβύη τα αποτελέσματα των επεμβάσεων είναι καταστροφικά χάος και αναρχία επικρατεί. οι πρόσφυγες προκειμένου να γλιτώσουν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον χάνουν τη ζωή τους στα νερά της μεσογείου. οι χώρες του νότου όπως η ελλάδα που έχουν υποστεί τα δεινά της οικονομικής κρίσης δέχονται κατά χιλιάδες σύριους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο. Σα ευχαριστώ κύριε Φουντούλη και τώρα για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Μίριαν Μον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την πληροφόρηση που μας δώσατε. Χαίρομαι που στις 9 Δεκεμβρίου ε, ξανάρχισε να δίνει ανθρωπιστική επιστηστική βοήθεια το πρόγραμμα σε πολλούς ήρους πρόσφυγες χάρη στην υποστήριξη και την ε, παγκόσμια και την ευρωπαϊκή τους επόμενους μήνες δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι θα βρούμε μπροστά μας την ίδια κατάσταση. Θα πρέπει να δεσμευτεί περισσότερο όλη η διεθνή κοινότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των σύρων προσφύγων τώρα που έρχεται και ο χειμώνας. Όπως είπατε Επίτροπε θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να αναζητούμε μια συνολική πολιτική λύση. Το πρώτο και το πιο επίγον βήμα είναι να μειωθεί η βία ε, για να επιτύχει αυτή η καινοτόμα πρόταση του ειδικού εμπεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Να υπάρχουν ε, διάδρομοι, ε, ζώνες ε, με παγωμένη σύραξη εχθροπραξία για να είναι δεδομένη η ασφάλεια και να μην εκτοπίζονται εκατοντάδες πολίτες και χιλιάδες. Χρειάζεται και πολιτική λύση όμως. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις μετριοπαθείς δυνάμεις στη Συρία. Έχουν χάσει ε, πρωταγωνισμό, έχουν αποδυναμωθεί γιατί τους επιτίθενται και οι κυβερνητικές ε, ένοπλες δυνάμεις και οι τρομοκράτες. Οι γειτονικέ χώρες και άλλοι διεθνείς παράγοντες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στις πλευρές για να τερματιστεί η σύραξη. Και τελειώνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνίστησε, όπω είπατε, Επίτροπε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και στην αναζήτηση πολιτική λύση τη σύγκρουση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ε, και ακολουθεί επόμενος ε, συνάδελφος ε, Φρουντσούλικα. μισή λεπτό. Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες αυτής ε, της δεκαετίας και δεν μοιάζει να τελειώνει. Ε, παραβιάζεται η ειρήνη, δολοφονούνται χιλιάδες άνθρωποι, καταστροφές σε αυτή τη χώρα, εκατομμύρια ανθρώπων που εκτοπίζονται ή καταφεύγουν στις ε, γειτονικέ χώρες. Παράλληλα όμως είναι απαραίτητο να προστατευτούν αυτοί οι πρόσφυγες και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα. 1,7 εκατομμύρια Σύρια, στην Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, ε, αυτοί που καλύπτονται από το ε, ανθρωπιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια τεράστια πρόκληση ε, στις ε, χώρες που άνοιξαν τις πόρτες τους στους πρόσφυγες δεν προσφέρουμε αλληλεγγύη και βοήθεια. Δεν θα πρέπει λοιπόν να διστάζουμε να αυξήσουμε τα κονδύλια μας λόγω της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία και στις όμορες χώρες. Έχουμε λοιπόν τους ιδιώτες δωρητές που βοήθησαν το παγκόσμιο πρόγραμμα πρόγραμμα το επισητιστικό, όμως αυτό δεν μπορεί να είναι η μόνιμη λύση. Παραμένει το θέμα στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται να τηρεί τις υποχρώσεις της. Οι πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να καταλήψουν τη χώρα τους, να ζουν σε καταφλισμούς, υποφέρουν από την πείνα και το κρύο, εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια. Η επιβίωση αυτών των ανθρώπων είναι καθοριστική σημασία και πρέπει να είναι δική μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε πολύ ε, συνάδελφε Φρουντσούλικα και ακολουθεί ε, για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος κ. Πράτσελ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τραγικό το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα αναγκάστηκε να σταματήσει τη βοήθειά του στη Συρία και επίσης είναι σαφές ότι στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται. Πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα και ισχύει αυτό και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κινητοποιηθούν περαιτέρω πόροι. Βεβαίως, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι χωρί την πολιτική άσκηση επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση ως έχει δεν θα είχε καν προκύψει. Όμως ε, εμείς ασχολούμεθα, εξακολουθούμε να ασχολούμεθα με τα συμπτώματα. Το θέμα δεν είναι μόνο να ανοίξουμε τα σύνορα και το πουγγί μας, αλλά ε, να φτάσουμε στα αίτια. Και έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα αραβικά κράτη. Αυτά όχι μόνο έχουν τα χρήματα, αλλά φέρουν και μια θρησκευτική ευθύνη, γιατί το βασικό πρόβλημα στη Συρία, το πρόβλημα είναι ο Ισλαμισμός ε, και όχι μόνο πρέπει να το θίγουμε το θέμα αυτό αλλά και να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Πχάτσελ για 1,5 λεπτό. Ακολουθεί ο συνάδελφος Νάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και την ευαισθησία την οποία επιδείξατε έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα ξανά, κάτι το οποίο είναι βασικό. Σας χειροκροτώ λοιπόν και το αναγνωρίζω. 5,5 εκατομμύρια θα προσθεθούν στα 18 που είχαν ήδη δοθεί. Ε, παραμένει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη σεβασμού των συμβιβαστικών λύσεων από πλευράς των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουν τον αγώνα τον οποίο δίδουν σε μόνιμη βάση με το Συμβούλιο θα πρέπει λοιπόν να ζητήσετε από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν υπόσχονται κάτι να το τηρούν. Πολύ ωραία. Η κυρία Αρναούτου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση των προσφύγων στην Συρία είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό και στην Ιορδανία και στο Λίβανο και στην Τουρκία να αναφερθώ στην κατάσταση των χριστιανών προσφύγων στον Λίβανο, ιδιαίτερα στο Τσάλε. Προέρχονται από τις επαρχίες του Όμς και του Άμα για να ξεφύγουν από τις διώξεις των ένοπλων ομάδων που έκαψαν τα σπίτια τους και που είχαν σαν σύνθημα των διώξεών τους να φύγουν οι χριστιανοί να πάνε στη Βηρητό και οι αλαουίτες να πάνε στον τάφο. Ε, δεν πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Οι τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους ε, βρήκαν καταφύγιο στην κοιλάδα της Μπέκα, ε, θεωρούνται πρόσφυγες και την χάνουν και πλέον εκτιμάτων οικονομικών. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να σταματήσει τις διακρίσεις εις βάρος των χριστιανών σύρων προσφύγων Κύριε Βαλενσιάνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Την περιέγραψαν την κατάσταση όλοι οι συνάδελφοι, είναι κρίσιμη. Ας φανταστούμε μια ευρωπαϊκή πόλη 1,7 εκατομμύριο. ας πούμε τη Βιέννη και ας ε, σκεφτούμε, αν φανταστούμε ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά είναι χωρίς ρούχα και χωρίς τροφή. Δεν θα είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν. Ε, πώς η κινητοποίηση θα δημιουργήσει μια τέτοια κρίση. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους λένε ότι δεν αντέχουν άλλο. Θα πρέπει να τρέχουν πίσω από τις κυβερνήσεις για να τις αναγκάσουν να ε, σεβαστούν τις υποχρεώσεις και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα ήδη κάνουμε. Και επίσης γνωρίζουμε ότι οι πιο πλούσιες χώρες θα πρέπει να μοιράσουν το βάρος για τις χώρες με τους ε, πρόσφυγες που έχουν εκατομμύρια, στο Λίβανο, η Ιορδανία, Τουρκία η δυνατότητα απορρόφησης των χωρών αυτών δεν είναι άπειρη ε, και εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε ε, απλοί παρατηρητές με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει οι ανεπτυγμένες χώρες, 130.000 Σύρους πρόσφυγες να υποδεχθούν, που είναι το 1 δέκατο των όσων υποδέχονται η Τουρκία ή ε, ο Λίβανος. Η Βραζιλία πήρε 1.500. Εμείς τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτή τη φορά λύθηκε η κατάσταση γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχετε την υποστήριξή μας ε, για να είμαστε στο πλευρό σα και αυτά τα πράγματα είναι τόσο απλά όσο και ε, απόλυτα είμαστε σε αυτό. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Ζητνάσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Από το 2011 Πάρα πολλοί υποφέρουν ε, στη Συρία λόγω της ένοπλης ε, σύραξης. Ε, εκατομμύρια αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις αιστείες τους και το 1 τρίτο αναγκάστηκε να καταφύγει σε γειτονικές χώρες. Αυτοί έχασαν τις αιστείες τους, τις δουλειές τους, αυτά που χρειάζεται κανείς για να επιβιώσει τρόφιμα και ζεστά ρούχα. Έχασαν και την αξιοπρέπειά τους. Το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα, στο οποίο συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, και εκτός από αυτή τη βοήθεια ε, θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ότι πρέπει να ξαναρχίσει το πρόγραμμα. Πολλοί Σύριοι πρόσφυγες βρέθηκαν σε πολύ πιο περίπλοκες θέσεις, σχέσεις διαβίωσης, αντιμετωπίζουν το κρύο. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να εμποδίσουμε το να υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι από το κρύο και την ασφάλεια. Νομίζω πρέπει να επιμείνουμε από αυτού. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστούμε πολύ ε, και δεν βλέπω στην αίθουσα της συνάλφου κυρία Τόγια. Κατόπιν τούτου ακολουθεί ε, κύριος Καν. Η βοήθεια πράγματι είναι απαραίτητη και είναι μεγάλη, μεγάλη ανακούφιση. Η διακοπή της χορήγησης τροφίμων μέσω του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος θα ήταν κάτι το τραγικό. Η αλήθεια είναι ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονται στα όρια τους λόγω του μεγέθους της κρίσης και απαιτούνται περαιτέρω πόροι για να λειτουργεί το σύστημα. Το θέμα δεν είναι να ζητάμε μόνο καλύτερη χρήση των πόρων οι οποίοι δεν είναι επαρκείς. Είναι πιο κρίσιμο να λύσουμε το πρόβλημα από τις ρίζες του. Συνδέεται βέβαια το μέγεθος της κρίσης με την διεθνή ανταπόκριση. Αν η διεθνή κοινότητα είχε ανταποκριθεί νωρίτερα απέναντι στη βιαιότητα του καθεστώτος Ασάντ, τότε η κατάσταση δεν θα είχε ξεφύγει και ακόμα και ε, το Ισλαμικό κράτος δεν θα είχε αποκτήσει ίσως τις διαστάσεις τις οποίες είχε σήμερα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση της περιοχής αυτής καλύπτοντας τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Είναι ηθική μας υποχρέωση. Ευχαριστώ κύριε Χάν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Λόπες. Πάει καιρός που η Συρία ζει ένα εμφύλιο πόλεμο με απολύτως αφόρητες και δραματικές συνέπειες. 200.000 είναι οι νεκροί, 11 εκατομμύρια οι Σύριοι που χρειάζονται σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια. Η μισή είναι παιδιά. 3,25 εκατομμύρια εκτοπισμένοι εκτός της Συρίας. 150.000 άνθρωποι έχουν ζητήσει άσυλο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και εκτός αυτού συστηματική ε, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιοπραγίες, βασανιστήρια, χρήση χημικών όπλων, αυτά είναι απολύτως αφόρητα. Και αυτή που είναι μάλλον η μεγαλύτερη τραγωδία σήμερα ε, στον κόσμο ανθρωπιστική, η δική μας απάντηση ήταν απολύτως ανεπαρκής, ανεπαρκέστατη. Γι' αυτό σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει τα εξής τέσσερα σαφέστατα μηνύματα. Πρώτον, ότι είναι έσχος το επιστημιστικό πρόγραμμα του ΕΕ που αφορά 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει ανασταλεί. Ακόμα και αυτό ήταν για μια εβδομάδα ε, πρόσκαιρο. Δεύτερο, ο Άσαντ δεν πρόκειται ποτέ να είναι τέρος μας. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένας παράγων εκεί για να βρεθεί μια πολιτική λύση στην περιοχή. Δεύτερο, τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό επίση. θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στην περιοχή και τέσσερα, πολύ σημαντικό επίση. θα πρέπει, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε τα 23 εκατομμύρια ευρώ πρόεδρος διακόπτη τον ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Λόπες. Και τώρα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Καπούτο. Ευχαριστώ. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τα Τρόφιμα προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες εκατομμυρίων σύρων που θίγονται από τον πόλεμο. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο αυτό θέμα. Ιδιαίτερα ξεχυμονιάζοντας μέσα σε πρόχειρες σκηνές πρέπει να βοηθήσουμε την οικονομία και των γειτονικών χωρών όπως η Αίγυπτος, η Ορδανία και κυρίως ο Λίβανος διότι η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί ε, έλλειψη σταθερότητας και τις γειτονικές χώρες. Πρέπει λοιπόν η διεθνής κοινότητα να ανταποκριθεί. Απαιτείται ε, επίσης να ξεκινήσει και το νέο μέσο στρατηγικής χρηματοδότησης ε, των προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Θέλω επίσης να συγχαρώ εδώ και την κυρία Μογκερίνη γιατί κάνει τεράστιες προσπάθειες για την επίλυση της ε, προβληματικής αυτής κατάστασης πιέζοντας και τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί και αυτή με τον δικό της τρόπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκάκελα για ένα λεπτό, Βάλει στο Κατσιά, η δεύτερη ομιλήτρια. Κυρία Σκάκελα, ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος πεινάει γιατί κράτη και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και εξακολουθούν να μην τις τηρούν. Και μετά τη νέα έκκληση του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που δεν ε, δίνουν τίποτα ενώ άλλα πάρα πολύ λίγα. Πρόκειται για πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία αυτοί. Και η σύραξη στη Συρία δεν είναι χτεσινή, ξαφνικά ξέσπασε χτες το βράδυ. Ούτε ο χειμώνα δεν είναι και καμιά τεράστια έκπληξη δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή να βρεθεί πολιτική λύση στη σύγκρουση. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Και πιστεύω ότι οι γειτονικέ χώρε τη Συρία κάνουν τεράστιε προσπάθειε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε για αύριο. Όποιο πεινάει σήμερα και είναι σε καταβλισμό προσφύγων δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να περιμένει. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Τώρα χρειάζεται δράση και να μην αφήσουμε μόνα του τα γειτονικά κράτη αλλά ούτε και του πρόσφυγες στη μοίρα του. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε και το χρόνο σα. Αυτοί οι δύο συνάδελφοι είχαν στήσει το λόγο για το Κασιά. Έξω όνομα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει επίτροπο κ. Σιλιανίδη. Παρακαλώ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να σε ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, ε, για όλα αυτά που είπατε και ευχαριστώ πολύ και για τα πολύ καλά λόγια που βρήκατε για μένα. Αισθάνομαι την υποστήριξή σας και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την υποστήριξη. Σε αυτή την τόσο δύσκολη δουλειά ε, που διεκπεραιώνεται και με τόσο δύσκολο τρόπο θα ήθελα να κλείσω την παρέμβασή μου με τρία ξεκάθαρα συμπεράσματα από τη σημερινή μας συζήτηση. Πρώτον, επαναλαμβάνω, η κρίση που συζητάμε σήμερα είναι χωρίς προηγούμενο. Τόσο σε επίπεδο ανθρωπιστικών συνεπειών για εκατομμύρια ανθρώπων και προφανώς και λόγω των ε, οικονομικών προεκτάσεων. Είναι μια κρίση που έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για μας, για την Ευρώπη. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση στον κανονικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς αυτή είναι μια αλήθεια. Όπως αναφέρατε, ε, μία είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αξιόπιστη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη συλλογική ευθύνη να βρούμε τα μέσα να το πετύχουμε αυτό. Και οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν επενδύσουμε επαρκή κονδύλια στην περιοχή, τότε οι συνέπειες ε, θα είναι ορατές και πολύ πέρα από την περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποκινούμε τα κράτη-μέλη για να βρούμε μια αποτελεσματική λύση στις ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της έχει ε, καταστεί ε, σημαντική στο να βρει την απάντηση. Είμαστε οι βασικότεροι δότες ε, και πρέπει να συνεχίσουμε να κατευθύνουμε αυτή την βοήθεια. Η ανθρωπιστική ε, αντίδραση δεν είναι κάτι που είναι ξεκομμένο. Πρόκειται για μια κρίση διαρκείας και απαιτεί μία ολοκληρωμένη απάντηση από κοινού ε, με οργανισμούς και εθνικές αρχές, αρμόδιες εθνικές αρχές. Ήδη συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας ε, για να εντάξουμε καλύτερα την ανθρωπιστική βοήθεια σε μια ολοκληρωμένη βοήθεια και χρειαζόμαστε να βρουμε τρόπους για να ενισχύσουμε την οικονομική βοήθεια που παρέχουμε. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτή η κρίση της ε, Συρίας, όπως αναφέρατε κι εσείς, απαιτεί πολιτική λύση. Δυστυχώς τα ανθρωπιστικά προβλήματα χρειάζονται πολιτικές λύσεις και ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα Επιγόντως πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να επιτύχουμε το στόχο μας. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξουμε τον κύριο Ντεμιστούρα, τον ε, ειδικό απεσταλμένο. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Σας ε, Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και πρέπει να σας πω ότι προσβλέπω στη συνέχιση της ε, συνεργασίας μεταξύ ημών σε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη και τώρα δίνω το λόγο με του Συμβουλίου στον κύριο Ντελαβέντοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση, να ευχαριστήσω και τον αρμόδιο επίτροπη για τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μας έδωσε. Δεν πρέπει να υπάρξει έλλειψη δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πρόκειται για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας από την αρχή της κρίσης ξεπερνάει τα 2,2 δις εκατομμύρια. Είμαστε από τους βασικούς χρηματοδότες και του Παγκόσμιου Ταμείου για τα Τρόφιμα. Η ανταπόκρισή μας στην τελευταία έκκληση ε, ε, απεδείχθη θα έλεγα η ανταπόκρισή μας ικανοποιητική. Οι πιστώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, να υπάρχει σωστός προγραμματισμός των προτεραιοτήτων, και είμαι βέβαιος ότι από κοινού θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους θέτουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση.